Να σας ανακοινώσω ότι από την ε, Ευρωπαϊκή Νοτική Αριστερά, Πράσινη Ευρωπαϊκή Αριστερά, το αίτημα από τον κύριο Γκουλιάνη, την, τον ορισμό του κύριου κύριο Γκουλιάνη ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται η τοποθέτηση. Πρώτο θέμα,